Καλημέρα κύριε Επίτροπε. Άρχεται η συνεδρίαση. Έχω μια ανακοίνωση να σας κάνω. Θα ήθελα να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι χθε οι αρχέ τη Αιθιοπία απελευθέρωσαν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Μερέρα Γκουντίνα μετά από κράτηση ενό έτου και πλέον. Ε, συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2016 στο αεροδρόμιο τη Αντίσα Μπέμπα επιστρέφοντας από τι Βρυξέλλε, όπου είχε συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε προηγούμενα ψηφίσματά του το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει την απελευθέρωσή του. Ε, ολόψυχα καλωσορίζουμε την απελευθέρωση απελευθέρωση αυτή και την απόφαση των αιθιοπικών αρχών. Είμαστε παγίω υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρώτο θέμα λοιπόν στην ημερήσια διάταξη είναι έκθεση του κυρίου Ντάντι. Εφαρμογή της οδηγίας των επαγγελματικών προσόντων και ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο